Συνεχίζει, ξανα, η συνεδρίασή μας. Τα αποτελέσματα του τρίτου γύρου για την εκλογή των αντιπρόεδρων είναι τα εξή. 656 μέλη εψήφισαν. Άκυρα ή λευκά 12. Έγκυρα 644. Οι επιμέρου υποψήφοι έχουν τον εξή αριθμό ψήφων. Ρομπέρτα ε, Αγγελίνη 274, Ιζαμπέλ Τιγό, 276 ψήφοι. Καμίσχη Μιχαλ Τόμα. 174, Σιλβάνα Κοχμερίν 186, Έντορα Μακμίλαν Σκοτ 294 ψήφοι. Μιγγέλ Αγχέλ Μαρτίνες Μαρτίνες 327 ψήφοι Δάκμα Ροτ 287 Λίμπο Ρούσεκ 278 Παλ Σμιτ 257 Αλέχο Βίνταλ Κβάτρας 308 ψήφοι Ταϊάννα Γόλις, 272 Κύριε Ράιναρ Βίλεν, 237 ψήφοι. Βάσει του τρίτου γύρου της ψηφοφορίας, σας αναγγείλω ότι έχουμε τώρα αντιπροέδρους, τον Μιχαήλ Αγγέλ Μαρτίνες Μαρτίνες, τον Βιντάλ Κάντρας, ε, Τάγμα Ροτ Πέντερ, Λίμπα Ρούτσεκ, Ιζαμπέλ Τουιγόν, Ρομπέρτα Αντζελίλη, Ταγιάννα Βόλης, Παλ Σμιτ, Μακμίλαν Σκότ, Ράινερ Βίλαντ και Σιλβάνα Κοχμερίνε. Θα ήθελα τώρα να συγχαρώ εγκαρδιότητα τους συναδέλφους που εξελέγησαν αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα συνεργαστούμε και η πρώτη μας συνεδρία του Προεδρείου δεν θα αργήσει να λάβει χώρα. Σύμφωνα με τον ε, κανόνα του κανονισμού 52, οι αντιπρόεδροι έχουν τη σειρά ανάλογα με τον αριθμό των ε, ψήφων που έλαβαν. Εάν υπάρχουν δύο που έχουν τον ίδιο αριθμό ψήφων, ο γερότερος είναι εκείνος που προηγείται. Διακόπτη συνεδρίαση μέχρι 9 της αύριο, το πρωί.